Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου. Παρακαλώ τους συναδέλφους που θέλουν να αποχωρήσουν να το πράξουν γρήγορα. Δεν ε, θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι οι ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο, γιατί θα ολοκληρωθεί η συνεδρίαση στις 2.30 και οι υπόλοιποι ομιλητές θα μπορέσουν να πάρουν το λόγο αύριο. Και άλλες δηλώσεις θα μπορούσαν να σταλούν και γραπτός. Να περάσουμε τώρα στην απαλλαγή 2013, Γενικός Προϋπολογισμός της Ένωσης. Η κυρία Λόπες Βερμέχο έχει το λόγο. Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Σήμερα είναι πολύ θλιβερή μέρα ε, για τους φίλους ε, του λαού της Σαχάρας ε, που έχει αντισταθεί με την ειρωνικό αγώνα τους κατά του βασιλείου του Μαροκοτοκοινοβουλίου ψήφισε με συντριπτική πλειοψηφία μια αναφορά στην διαχείριση